Για να ξαναξεκινήσουμε, να δούμε λοιπόν και τα χθεσινά πρακτικά και τα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν και τα οποία είναι στη διάθεσή σας. Κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο για κάτι από τα πρακτικά. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να εγκρίνουμε ε, τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης στην οποία μόλις αναφέρθηκα. Το πρώτο σημείο που έχουμε στην ε, ημερήσια διάταξη